Καλημέρα σας. Θα αρχίσουμε με ορισμένες ανακοινώσεις. Σε σχέση με τους συντονιστές, δηλαδή τις αποφάσεις που λάβαμε κατά τη διάρκεια των, της συνεδρίασης των συντονιστών. Σας υπενθυμίζω καταρχήν ότι η συνεδρίασή μας, η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, τη συνεδρίαση αυτή μπορείτε να, μπορεί να ε, την παρακολουθήσει κανείς και από το διαδίκτυο. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ιθογένεια ορίστηκε η κυρία Γκουρμάη υπεύθυνοι, γιατί υπάρχει και ένα αίτημα από το ΔΕΚ για την τροποποίηση του καθεστώτος και διορίστηκε ως εισηγητής για γνωμοδότηση ο κύριος Μέσερ Σμιτ σε σχέση με το δικαιοδοτικό σύστημα με συγχωρείτε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας η σοσιαλιστική ομάδα θα ορίσει τον εισηγητή. Στη συνέχεια αποφασίσαμε στις 9 και 10 Νοεμβρίου εδώ στις Βρυξέλλες να ακούσουμε εμπειρογνώμονες από το Παρατηρητήριο για τη Δημοκρατία σε σχέση με τις μελέτες που έχει αναλάβει το παρατηρητήριο αυτό για θέματα δημοκρατίας στην Ευρώπη. Τέλος, εξετάσαμε το αίτημα της κυρίας Γκουρμάη να προωθήσουμε μία συζήτηση στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για το, μια συζήτηση για το Ουγγρικό Σύνταγμα. Θα ορίσουμε την ημερομηνία, δεν έχει ακόμα οριστεί και θα ακούσουμε έναν μόνο εμπειρογνώμονα. Είναι ο δόκτωρ Κουχουρέλη, όπως όρισε η κυρία ε, Γκουρμάη και θα αναφερθούμε μόνο στην Ευρωπαϊκή Ρήτρα και τις επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Συντάγματος σε σχέση με τα θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η, η ημερομηνία θα οριστεί λίγο αργότερα για τις 5 ή 10 Οκτωβρίου. Άλλες ανακοινώσεις. Περνάμε στις άλλες ανακοινώσεις. διακοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας συμμετείχα στη συνεδρίαση της ΑΦΕΤ της 22ης Ιουνίου και ένα σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια Μεταγενέστερα όπου εκφράστηκε μία επιφύλαξη ως προς την ενδεχόμενη, μία ενδεχόμενη πρόταση ψηφοφορίας επί του θέματος χωρίς να έχει γίνει διαβούλευση με την ΑΦΚΟ. Γιατί όπως ξέρετε το θέμα αυτό σε σχέση με τα, και με τα εθνικά κοινοβούλια αφορά την ε, Επιτροπή μας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τις διακοινοβουλευτικές σχέσεις και το θέμα αυτό δεν αφορά αποκλειστικά το Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό έκρινα, κρίναμε ότι η ΑΦΕΤ θα πρέπει να αποφανθεί έτσι ώστε να επηρεαστεί και το Συμβούλιο. Το άρθρο 9 του πρωτοκόλου υπαριθμών 1 αφορά την ε, αποτελεσματική διακοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ δηλαδή εθνικών κοινοβουλίων και ευρωπαϊκού. Η πρόταση ψηφίσματος εγκρίθηκε, έκρινα σκόπιμο να σας μιλήσω για τις επιφυλάξεις, τις μεταγενέστερες επιφυλάξεις. Στις 30 Ιουνίου η Επιτροπή οργάνωσε μία συνεδρίαση με εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την πρωτοβουλία για τους πολίτες. Ζητήθηκε με βάση την Συμφωνία Πλαίσιο από την Επιτροπή να καλέσει και εμπειρογνώμονες από τη δική μας Επιτροπή. Άρα, σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών συμμετείχαν και μέλη της δικής μας γραμματείας στη συνάντηση αυτή της 30ης Ιουνίου. και διαφέρει η προετοιμασία της εφαρμογής του κανονισμού από κράτος σε κράτος, ιδιαίτερα σε σχέση με την ηλεκτρονική ψηφοφορία που ορισμένα κράτη δεν μπορούν επί του παρόντος να διοργανώσουν. Δεν διαθέτουν δηλαδή τα κατάλληλα μέσα για να προετοιμάσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουν στο σημείο να την διαθέτουν. Ως προς τον κώδικα συμπεριφοράς της 5 Ιουλίου, πρόεδρος Μπούζεκ σε μια άτυπη συνεδρίαση της συνεδρίασής μας μίλησε για τον κώδικα συμπεριφοράς της ομάδας εργασίας. Εμείς όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε με την τροποποίηση του κανονισμού δύναμη του άρθρου 212 και θα ορίσουμε, θα διορίσουμε και εισηγητή. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, περνάμε στην ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν τώρα στις ε, ψηφοφορίες σε σχέση με την ερμηνεία του άρθρου 51 του κανονισμού μέσα στα πλαίσια των ε, διεθνών ε, συμβάσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελε ε, ο εισηγητής να προσθέσει κάτι ή όχι. Δεν ζητά το λόγο, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα την φόρμουλα αυτή της ερμηνείας που πρότεινε ο David Μάρτιν σε σχέση με την ερμηνεία του άρθρου 51 του κανονισμού, δηλαδή το σημείο 8. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ της πρότασης κατά αποχές εγκρίνεται. Ομόφωνα η ερμηνεία του άρθρου 51. Η δεύτερη ψηφοφορία αφορά τις μονομερείς δηλώσεις στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Ήδη έγινε συζήτηση για τις τροπολογίες, δεν ξέρω κατά πόσο ο εισηγητής θα ήθελε κάτι να προσθέσει. Uh, ο εισηγητής, ο κύριος Τσαρκόφσκι. Ε, σε σχέση με την 7 έχω μία προφορική τροπολογία. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε μέχρι την ε, τροπολογία 7, όπου θα σας υποβάλω μία προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν το έγγραφο για τις μονομερείς δηλώσεις που εγγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Ψηφίζουμε το άρθρο 4, μάλλον με συγχωρείτε, την τροπολογία 4. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5. Παράγραφος 1α. Νέα παράγραφος γκουρμάι Υπέρ. Κατά. απορρίπτεται εμφανώς. 6 στην παράγραφο 1α, νέα παράγραφο, DAF υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7. Τροπολογία 7 και ακούμε τον εισηγητή. Λάβαμε μία γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο σαφείς στο κείμενο της έκθεσης, γι' αυτό να πούμε σε σχέση με τις δηλώσεις των κρατών μελών, έτσι ώστε να μην δημοσιεύονται στην σειρά L της επίσημης εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αυτή είναι η προφορική. Ψηφίζουμε την τροπολογία 7 με την προφορική Ποιοι είναι υπέρ της 7 τροποποιημένης, ούτως τροποποιημένης, κατά 2. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Σασκόφσκι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόκειται για την αιτιολογική σκέψη ε. 2. Ιμπράσας υπέρ, κατά Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Πάξας. Α, όχι, καταπίπτει. Όχι, όχι, πρέπει να ψηφιστεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία του σχεδίου όπως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελευταία ψηφοφορία αφορά την ερμηνεία στο άρθρο 192. Το άρθρο 192. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε για τη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων βουλευτών στις συνεδριάσεις των συντονιστών να είναι το τελευταίο θέμα. Και αυτή η γνωμοδότηση διατυπώθηκε υπό μορφή επιστολής και ανακύπτει από το γεγονός ότι δύο επιτροπές ζήτησαν στη συνεδριάση των συντονιστών να μπορούν να συμμετέχουν και οι μη εγγεγραμμένοι. Μάλλον εκπρόσωποι των μη, ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων. Και υπάρχει και η επιστολή. Vabbè, ε. poi Υπάρχει λοιπόν ένα Έτοιμα. Με συγχωρείτε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Υπάρχει ένα αίτημα έτσι ώστε να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων στη συνεδριάση των συντονιστών. Υπάρχει λοιπόν αυτό το Έτοιμα. αλλά επειδή δεν ε, προβλέπει κάτι τέτοιο ο κανονισμός θα πρέπει να αποφανθούμε. έτσι ώστε ένας εκπρόσωπος από τους μη εγγεγραμμένους να συμμετέχει συνεδριάσει των συντονιστών. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αποφανθούμε και δεχτήκαμε στη συνεδριάση των συντονιστών να μην, να μην συμμετέχει ένας μη εγγεγραμμένος με δικαίωμα ψήφου, αλλά ένα μέλος της γραμματείας των μη εγγεγραμμένων που μετά ενημερώνει τους μη εγγεγραμμένους για τα τεκτενόμενα στις συνεδριάσεις. Γι' αυτό εμείς κρίναμε ότι θα πρέπει να συμβαδίσουμε με, τις, ε, με αυτά που ε, αναφέρουν οι περισσότερες ε, επιτροπές, δηλαδή η πλειοψηφία των επιτροπών, έτσι ώστε να μην συμμετέχει ένας μη εγγεγραμμένος, αλλά να μπορεί να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες από ένα μέλος της γραμματείας. Αυτό θα ήθελα να ψηφίσουμε. Θα ήθελε κάποιος να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Κλάης, σήμερα ήρθε στην Επιτροπή αυτή ε, γιατί δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ούτε το τακτικό μέλος ούτε το αναπληρωματικό. Θέλω να παρακολουθώ την κατάσταση εκ μέρου των μη εγγεγραμμένων. Έχουμε πρόβλημα πρακτικό γιατί δεν μπορούμε να συμμετέχουμε συνεδριάσεις των συντονιστών. Γνωρίζετε ότι οι εκθέσεις, για παράδειγμα, μοιράζονται στις συνεδριάσεις των συντονιστών. Εκεί ορίζονται οι συγγητές ε, σε κάθε έκθεση ας πούμε και οι μη εγγεγραμμένοι έχουν δικαίωμα να αναλαμβάνουν εκθέσεις όπως όλα τα άλλα μέλη του Κοινοβουλίου και να είναι συγγητές. Λοιπόν, τίθεται το πρακτικό ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν για όνομα του Θεού, ένα μη εγγεγραμμένο μέλος να οριστεί εισηγητής εφόσον απουσιάζει στην συνεδρία των συντονιστών όπου αποφασίζεται ποιος θα είναι ο εισηγητής και οι εκθέσεις είναι μια κατάσταση που υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από επιτροπή σε επιτροπή. Σε ορισμένες επιτροπές, ε, καμιά φορά επέτρεπα να είναι παρόντες και μία εγγεγραμμένη ή τουλάχιστον ε, ε, από τη γραμματεία, από το προσωπικό μας και έπαιρναν καμιά φορά και καμιά έκθεση. Σε άλλες επιτροπές ε, είναι τελείως αδύνατο με οποιοδήποτε τρόπο να έχουμε εκπροσώπηση. Υπάρχουν επιτροπές με πόντους, υπάρχουν επιτροπές χωρίς point system και ε, σε άλλες επιτροπές παίρνουν πόντους οι μία γεγραμμένοι, σε άλλες δεν παίρνουν. Είναι μια τεράστια αδικία μεταξύ των βουλευτών αλλά και μεταξύ των διαφόρων επιτροπών αυτή που επικρατεί. Στο ίδιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τα άλλα και θα ήθελα να κάνω την πρακτική ερώτηση. Ποια δυνατότητα βλέπετε εσείς και τι προβλέπετε για τους μη εγγεγραμμένους για να παίρνουν εκθέσεις, να γίνονται και εισηγητές ε, όταν δεν τους επιτρέπεται η παρουσία στη συνεδρίαση των συντονιστών. Με άλλα λόγια, στην καλύτερη περίπτωση ενημερώνονται, λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων εκ των υστέρων. Δηλαδή κάθε φορά είναι αδύνατο να πάρεις έκθεση αν είσαι μη εγγεγραμμένος. Και είναι και άλλα θέματα ε, περιορίζομαι μόνο στην ιδιότητα του εισηγητή. Υπάρχουν και άλλα πρακτικά προβλήματα όμως, όπου δεν μπορούμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί, όπως άλλα μέλη του Κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε μια πολιτική ομάδα. Ερωτώ, ποια διαδικασία προβλέπετε εσείς τώρα για ένα μέλος του Κοινοβουλίου που δεν είναι γεγραμμένο σε πολιτική ομάδα για να πάρει έκθεση. Το πρόβλημά μου είναι το εξή σα. δούμε τι θα πούν και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, αλλά εγώ πρέπει πρώτο μου μέλημα, πρωταρχικό μου μέλημα, ε, είναι να εφαρμόσω τον κανονισμό. Ο κανονισμός άλλαξε από την έκθεση Corbett και αναφέρεται ότι ενδεχομένως ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων θα μπορούσε να συμμετέχει στην συνεδρία των συντονιστών. Η έκθεση Κόρμπετ άλλαξε τα δεδομένα και εγκρίθηκε η έκθεση Κόρμπετ όπως γνωρίζετε από την Ολομέλεια. Άρα οι μη εγγεγραμμένοι δεν μπορούν να συμμετέχουν. Εγώ δεν έχω την εξουσία να αλλάξω αποφάσεις που έχουν ήδη λεφτεί. Γνωρίζω βέβαια ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Σας ρωτώ λοιπόν πώς μπορούμε να, να, το κάνουμε έτσι ώστε και οι μη εγγεγραμμένοι να μπορούν να αναλάβουν μια έκθεση. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι το θέμα προ... τα θέματα προσυζήτησης τους συντονιστές μπορούν να γνωστοποιηθούν στους μη εγγεγραμμένους ήδη από πριν. Άρα μπορούν γραπτός να ζητήσουν την ανάληψη μιας έκθεσης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Τώρα, η φυσική παρουσία στους συντονιστές των μη εγγεγραμμένων δεν προβλέπεται. Και αυτό δεν είναι και αποφασιστική σημασία όταν ψηφίζουμε, ειδικά όταν πρόκειται για κάτι το συνενετικό. Αποφασιστική σημασία είναι να, να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον τους. Και δεν νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη αυτό το αίτημα. Ο κύριος Ντάφ ζήτησε το λόγο. Ζόντεργκαρτ, Πριν. Ευχαριστώ αναγνωρίζω πολύ καλά, καταλαβαίνω την ε, επιχειρηματολογία και γνωρίζω τι νόημα έχει και η έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, ε, ο λόγος που προβάλλεται αυτό το αίτημα είναι ο εξής. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πολύ ε, δύσκολη η σύσταση πολιτικών ομάδων και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια μεγάλη ομάδα η οποία βρίσκεται εκτός πολιτικών ομάδων. Αυτή η συζήτηση ανέκυψε κατά την τελευταία θητεία, όπου οι δύο μεγάλες ομάδες είχαν αποφασίσει να καταστήσουν πιο, αυστηρούς, πιο αυστηρό το πλαίσιο λειτουργίας των πολιτικών ομάδων. Δηλαδή είναι πιο δύσκολη η σύσταση πολιτικών ομάδων και πολλοί βουλευτές βρέθηκαν εκτός πολιτικών ομάδων. Αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει, είναι πολύ σοβαρό. Αυτό είναι το πρόβλημα ουσίας που διέπει αυτή τη συζήτηση. Όπως σας είπα, θα ήθελα να καταβάλουμε μια προσπάθεια ως Επιτροπή να προβάλλουμε αυτή τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε ο κανονισμός να είναι πιο ολοκληρωμένος και να μπορούν και οι μη εγγεγραμμένοι να έχουν αυτό το δικαίωμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νταφ, θα ήθελα όμως πληροφοριακά να σας υπενθυμίσω το εξής, κάτι το οποίο δεν αναφέραμε πριν. Η συνεδρίαση των συντονιστών δεν έχει δικαίωμα λήψης αποφάσεων, δηλαδή προβάλλει προτάσεις. Όταν πρόκειται για εκθέσεις, οι συντονιστές δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις. Πολλές φορές ε, εξουσιοδότηση μπορούν να λάβουν μία απόφαση. Άρα η ίδια Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις. Άρα υπ' αυτή την έννοια οι μη εγγεγραμμένοι μπορούν να προβάλλουν μία γνώμη επί του θέματος. Ο κύριος Ντάφη έχει το λόγο. Συμφωνώ Πρόεδρε, με την ε, δική σας ε, ε, ερμηνεία σχετικά με τη λειτουργία των συνεδριάσεων των συντονιστών, το ρόλο των συντονιστών. Εμείς είμαστε συντονιστές και εκπροσωπούμε πολιτικές ομάδες που απαρτίζονται από μέλη που έχουν κάποια πολιτική συγγένεια. Συμφωνώ με τον κύριο Σόντεγκα βεβαίω. πως είναι δύσκολο ή δύσκολα τα πράγματα Αφήστε που έχει παραμείνει σταθερός ο αριθμός των μη εγγεγραμμένων για διάφορες διαδοχικές θητείες σε σχέση με τους βουλευτές που προσχωρούν σε κάποια πολιτική ομάδα. Συμφωνώ βεβαίως με αυτό αυτά που μας είπε ο κύριος Μπρόνς, αν επιθυμεί να γίνει συγητής, θα έπρεπε να ενημερώσει τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής και η ίδια η επιτροπή θα αποφασίσει. Μέχρι στιγμής ο κύριος Μπρόνς δεν έχει εκφράσει καμία επιθυμία να υπηρετήσει την Επιτροπή με την ιδιότητα του εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σέφνερ. Εδώ βρισκόμαστε όλοι γιατί μας έχουν στείλει πολίτες που μας έχουν ψηφίσει ε, βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως βουλευτές έχουμε και κάποια δικαιώματα και κάποιες υποχρεώσεις. Τελείως ανεξάρτητα, δηλαδή, ε, καταρχήν από τη συμμετοχή σε πολιτικές ομάδες. Το ερώτημα το βρίσκω πάρα πολύ θεμητό. Πώς μπορεί ένας βουλευτής που δεν είναι μέλος μιας πολιτικής ομάδας να ασκεί τα δικαιώματά του όσο και τις υποχρεώσεις του πλήρως ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτόμαστε και το να βάλουμε υπόψη στις αποφάσεις που παίρνουμε. Τώρα άλλο θέμα είναι η συνεδριάση των συντονιστών. Οι συντονιστές εκπροσωπούν όντω πολιτικές ομάδες και εξ αυτού ε, έχουν μια ιδιαίτερη ε, νομιμοποίηση που βασίζεται στο κανονισμό. Και εκείνοι που δεν θέλουν ή δεν μπορούν ε, να συστήσουν πολιτική ομάδα δεν εντάσσονται. Λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε μια λύση και τα δύο θέματα είναι πολύ σημαντικά από πλευρά συνταγματική. Θα μπορούσα να φανταστώ εδώ να πάμε ακόμα παραπέρα από αυτό που προτείνει ε, αυτό που είπε ο Πρόεδρος, δηλαδή ένας εκπρόσωπος των ε, μη εγγεγραμμένων βουλευτών να επιτρέπεται να συμμετέχει συνεδρία των συντονιστών, αλλά ευθύ εξ αρχή να έχει διακριτό ρόλο. Er δεν είναι συντονιστή γιατί δεν εκπροσωπεί πολιτική ομάδα, αλλά δεν θεωρώ απαραίτητο ή υποχρεωτικό να είναι βοηθός ή, ή συνεργάτης και όχι μέλος παρευρισκόμενος. Αυτό απέχει λίγο ω ερμηνεία από τι μέχρι τώρα ερμηνείε που δίνει το Κοινοβούλιο και το λέω και εξ ονόματο τη ομάδα μου. Κατά τα άλλα τα ίδια ε, υποστήριξα και στη Γερμανική Βουλή, στην Bundestag, έκαναν την ίδια πρόταση και τότε οι σοσιαλδημοκράτες και συντηρητικοί το απέρριψαν. Και τι έγινε, πήγαν στο συνταγματικό δικαστήριο οι μη εγγεγραμμένοι και το συνταγματικό δικαστήριο τους δικαίωσε και επέβαλε τη συμμετοχή τους ε, στα κοινοβουλευτικά πράγματα το κοινοβούλιο δεν θα βλάψει τον εαυτό του αν έχει ε, ένα οργανωμένο τρόπο να ενημερώνονται, να συμμετέχουν και όπου έχουν το δικαίωμα ε, να ε, επιδρούν και στη συνεδρίαση τέτοια μέλη που δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα. Λοιπόν, θεωρώ σωστό αυτό που τώρα προτάθηκε ενημέρωση, ε, ημερήσια διάταξη, παρατηρητές να μπορούν να στέλνουν, όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά εγώ θα έκανα και το επόμενο βήμα και θα έλεγα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά βοηθός ενός βουλευτού, μπορεί να είναι και βουλευτής. Ο οποίο όμω βουλευτή δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με του υπολείπου συντονιστέ. Ε, δεν μπορεί να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. κύριος Κλάης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω και βλέπω ότι υπάρχει κατανόηση για την κατάσταση των μη εγγεγραμμένων. Γιατί με είναι καλό πράγμα αυτό. Ε, πάντως στο μέλλον υπάρχει δυνατότητα και φαίνεται αυτό να βρεθεί κάποια λύση. Δεν έχω πιστεί τελείως από ε, αυτά που είπατε πρόεδρε προσπαθώντας να με καθησυχάσετε γιατί πρακτικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενημερωνόμαστε εκ των προτέρων για το ποιες εκθέσεις θα μοιραστούν σε μια τέτοια συνεδρία των συντονιστών. Διότι στην Επιτροπή Ελευθεριών που είμαι εγώ μέλος παίρνονται οι αποφάσεις κανονικά στη συνεδρίαση των συντονιστών για το ποιο θα κάνει την έκθεση. Και μας, μας ενημερώνουν στη συνέχεια στην Επιτροπή κατόπιν εορτή. Τι να το κάνω. Και ποτέ δεν αμφισβητεί κανείς απόφαση των συντονιστών, ούτε την προσβάλλει. Οπότε θα μπορούσαμε να βρούμε μια ενδιάμεση λύση, κατά αναλογία με τη διάσκεψη των Προέδρων, να έχουμε έναν εκπρόσωπο των μη εγγεγραμμένων που να μην έχει τα ίδια δικαιώματα. Εντάξει, συμφωνώ. Οι μη εγγεγραμμένοι, το ξέρω, δεν είναι ομοιογενής πολιτική ομάδα, ούτε μπορούν να εξισωθούν σε καμία περίπτωση με μια πολιτική ομάδα. Συμφωνώ. Αλλά με κάποιο τρόπο να έχουμε δικαίωμα να ακουγόμαστε στους συντονιστές. Αυτό τώρα που προβλέπετε να επιτρέπετε παρουσία κάποιου υπαλλήλου στη συνεδρία των συντονιστών, καταλαβαίνετε ότι ένας υπάλληλος ή ένας βοηθός ε, δεν θα έχει καν δικαίωμα λόγου. Ε, ε, θα είναι απλώς παρατηρητής. Οπότε δεν θα μπορούμε ποτέ τα μελήματά μας, τις ανησυχίες να σας τα διαβιβάζουμε σε μια τέτοια συνεδρίαση και πάντα θα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις στην ε, δική μου γνωμοδότηση. Άρα θα υπάρξει η διευκρίνηση ότι οι μη εγγεγραμμένοι μπορούν να ζητήσουν να αναλάβουν μία έκθεση από τον Πρόεδρο. Και η απόφαση θα ληφθεί από τη... λαμβάνεται από την Επιτροπή και όχι από τους συντονιστές έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει η εγγύηση ε, της παρουσίας ενός εκπροσώπου από τη γραμματεία. Αλλά ως προς έναν βουλευτή μη εγγεγραμμένο δεν μπορεί εκείνος να εκπροσωπήσει τους πάντες. Γι' αυτό η γραμματεία θα πρέπει να ενημερώνει τους μη εγγεγραμμένους. Θα ήθελα να ψηφίσουμε τη δική μου γνωμοδότηση. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ της γνωμοδότησής μου. Κατά. Αποχές. Έχουμε τέσσερις αποχές. Τέσσερις αποχές. Άρα έχουμε τελειώσει με τις ψηφοφορίες και πριν περάσουμε στο τελευταίο θα ήθελα να καλωσορίσουμε την κυρία Έπεριν Λίν Ρέγνερ, η οποία συμμετέχει στις εργασίες μας, αν και αναπληρωματικό μέλος. Πρόκειται για μία συνάδελφο η οποία βρίσκεται, είναι πάντα παρούσα στις εργασίες και παρά το γεγονός ότι είναι αναπληρωματικό μέλος θα μπορέσει να συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες μας. Σας εύχομαι λοιπόν μια πολύ καλή συνεργασία. Ας περάσουμε στο τελευταίο θέμα που είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτών. Ο συνάδελφος ε, Τσασκόφσκι ορίστηκε ε, εισηγητής και είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων χωρίς έγγραφο. Θα ήθελα λοιπόν ο συνάδελφος Τσασκόφσκι να μας ε, εκφράσει την άποψή του, δηλαδή τις υποδείξεις που θα ενταχθούν στη συνέχεια στην έκθεση Μπερές. Συνάδελφοι, θα μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο από θεσμικής πλευράς. You have my opinion in front of you. Έχετε τη γνωμοδότησή μου Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό καθ' αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο, διότι Υπάρχει το θέμα των νομικών μηχανισμών ε, δευτερογενούς δικαίου και κατά πόσο είναι αποτελεσματική και επίσης διατίθεται θέμα ε, νομικής ασφάλειας. Αφήστε που μιλώντας για την οικονομική διακυβέρνηση, πέρα από το εξάμεινο υπάρχουν μεγάλες παρανοήσεις και θα πρέπει η Επιτροπή μας ε, κάπως να χειριστεί το θέμα. Πρώτον, υπάρχουν διάφορα δεσμευτικά και μη εργαλεία τα οποία προσπαθούμε να επισημοποιήσουμε. Δεύτερον, δεν είναι διόλου σαφές ε, δηλαδή ε, δεν ξέρουμε πώς να αποδοθούν οι ευθύνες, ποιος φέρει ποια ευθύνη. Εδώ μιλάμε για μέλη της ζώνης του ευρώ, του συμφώνου EuroSyn ε, και υπάρχει και η σύγχυση σε σχέση με τις ευθύνες σε επίπεδο κράτων μελών επίσης. Θα θέλαμε να διευρύνουμε τη γνωμοδότηση, να μην ασχοληθούμε μόνο με το ευρωπαϊκό εξάμεινο, να εκφράσουμε την ανησυχία μας για αυτό που σας είπα, το θέμα της νομικής ασφάλειας και το θέμα ε, της λογοδοσίας των ευθυνών. Και γι' αυτό συμπεριέλαβα αυτή την παράγραφο. Ο στόχος ε, της ε, γνωμοδότησης είναι όχι μόνο να εκφράσουμε τους ενδιασμούς μας σχετικά με την νομική ασφάλεια, αλλά το πιο σημαντικό είναι να επισημοποιήσουμε την ε, συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2010, συγκεκριμένα ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αφορά σε όλα τα κράτη-μέλη, τα 27 κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ε, ως προς το νομικό σύστημα διότι υπάρχουν μηχανισμοί ε, συντονιστικοί δευτερογενούς δικαίου και είδαμε με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού συνθήκη της Λισαβόνας ότι τέτοιου είδους μηχανισμοί δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Επίσης, ε, τονίζω ότι κατά την επισημοποίηση πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι θεσπίζουμε εργαλεία που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ως προς την νομική φύση τους. Προφανέστατα το πλέον σημαντικό για μας δεν είναι μόνο να προβλεφθούν αυτά στην ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με τρόπο ώστε να διατηρηθεί η εισαγωγικά κοινοτική μέθοδος, κυρίως σε σχέση με την, ε, ε, το δικαίωμα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εποπτική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η προσέγγιση της περιβάλλοντος περές παρεπιπτόντος συνάδει με αυτό, δηλαδή προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και στην περίοδο της εποπτείας κατά την εφαρμογή της διαδικασίας. Οπότε ε, παρατηρούμε μια διάσταση απόψεων σχετικά με την προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσουμε και έγινε συζήτηση αν χρειάζεται διαθεσμική συμφωνία ή αν επαρκεί ένας κανονισμός ή αν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική οδός, ώστε να σωματώσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο στην ένωμη τάξη της Ένωσης. Εκρεμεί ακόμη το ζήτημα, παρότι ε, εγώ προσωπικά προτιμώ να χρησιμοποιήσουμε ένα κανονισμό και όχι να καταλήξουμε σε διαθεσμική συμφωνία. Η Πρεβάνσε Μπερές νομίζω εξετάζει το ενδεχόμενο να ακολουθήσουμε ακόμη και μια τρίτη εναλλακτική λύση για να ρυθμίσουμε το ζήτημα. Κατόπιν μιλάμε για το ρόλο του, Εθνικού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εντελεχώ στην παράγραφο 6 μιλάμε για την ε, δημογραφική νομιμοποίηση ε, και ότι πρέπει να εμπλέκεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και κυρίω ω προ τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται, ε, ω προ την αξιολόγηση κατά το πέρασε του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα ήθελα να πω ότι εκκρεμεί το ζήτημα διότι θελημένα μάλλον, διότι ε, ακούστηκαν ιδέες σχετικά με αυτές τις μικτές ε, διασκέψεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών αλλά θα το αφήσουμε ανοιχτό το ζήτημα γιατί παρακολουθούμε και τις διαπραγματεύσεις για το πακέτο των έξι οδηγιών για την οικονομική διακυβέρνηση. Ε, ε, τώρα με, λειτουργούμε βάσει χρονοδιαγράμματος και πρέπει να, το, να έχουμε επίγνωση ε, αυτού. Η έκβαση των διαπραγματεύσεων για το πακέτο των ΕΚΣ θα επηρεάσει και τη θέση μας εδώ. Γνωρίζω ότι θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις το Σεπτέμβρη και για το ευρωπαϊκό εξάμεινο κάποιες γενικές διατάξεις συμπεριλαμβάνονται ήδη σε ένα από τα σχέδια κανονισμού. Ε, και... Όπως ε, είπε και η Περβάνς ε, ε, Μπερές, ο στόχος είναι να περάσει από την Επιτροπή και από την Ολομέλεια σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία. Προφανέστατα είναι συναφή τα ζητήματα. Δεν πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού. Αλλά καθότι δυστυχώς ανεβλήθησαν αυτές οι διαπραγματεύσεις, δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων γιατί είναι ελέγχητα τα ζητήματα. Θα ε, παρακολουθήσουμε λοιπόν τις εξελίξεις αν δεν θέλουμε να είναι ε, άσκοπο ουσιαστικά το, ε, το σχέδιό μας. Και όπως σας είπα, μέσα στην έκθεση παραμένω να αφήσω για τη σχέση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτά για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η Επιτροπή μας ε, είναι στην αρμοδιότητα μάλλον της Επιτροπής μας να εκφράσει τουλάχιστον τις ανησυχίες σε σχέση με αυτά τα θέματα της νομικής ασάφειας κατόπιν ε, επισημοποίηση της όλης ε, διαδικασίας θα πρέπει να προαγάγουμε τη διαδικασία και να προσδιορίσουμε με ποιο τρόπο ακριβώ, δηλαδή να εκφράσουμε την προτίμησή μα και τρίτο και τελευταίο για να διατηρηθεί η κοινοτική μέθοδο και οι αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να κινηθούμε με πυγμή προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, όλα αυτά, ξαναλέω, η θελημένα άφησα σαφή δύο ζητήματα μέσα στην έκθεση γιατί όπω σα εξήγησα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τη εξελίξη, διαπραγματεύσει για το πακέτο των έξω για την οικονομική διακυβέρνηση Ευελπιστούμε πάντως να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση, να καταλήξουν μάλλον σε συμβαστική λύση και μετά ε, ευελπιστούμε ότι θα μπορούμε να γίνουμε και εμείς πιο συγκεκριμένοι. Αυτά και περιμένω τα σχόλιά σας ε, για το σχέδιο και για όλες αυτές τις παρατηρήσεις που έκανα παρουσιάζοντας το σχέδιο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Αρχίζει η συζήτηση. Ο κύριος Μπολτιέρη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσασκόφσκι για αυτό το προσχέδιο γνωμοδότησης το οποίο ασχολείται με τις βασικότερες ε, θεσμικές επιπλοκές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα πρέπει να αποσαφινιστούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει ένα ανεπαρκές και κατά προσέγγιση νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να προβούμε σε ένα συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της Ένωσης και των κρατών μελών στα πλαίσια της συμμετοχής του στην Ένωση, διότι όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αφορά την αναθεώρηση του κώδικα συμπεριφοράς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Άρα το βασικότερο θέμα για τη δική μας Επιτροπή έγκυται στο να ορίσουμε κάπως καλύτερα, να οριοθετήσουμε το εξάμεινο με αυτή την γνώμη, τη γνωμοδότηση. Νομίζω λοιπόν ότι το σκεπτικό μας ίσως οδηγήσει σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που προτείνει ο εισηγητής. Ο εισηγητής προτείνει να δώσουμε επίσημο χαρακτήρα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με βάση το άρθρο 121 σημείο 6 μέσα στα πλαίσια του κανονισμού που εποπτεύει και συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές, δηλαδή τον κανονισμό του 97 που έχει αναθεωρηθεί από την έκθεση wortmann κόλ, Άρα έχουμε να βασιστούμε σε έναν κανονισμό και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να το εντάξουμε σε αυτό το συγκεκριμένο κανονισμό που αποτελεί ένα από τα πακέτα της διακυβέρνησης που με τη σειρά του αποτελεί μία από τις ε, πτυχές της στρατηγικής 2020. Ε, κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι συρρυκνώνουμε το όλο πλαίσιο Δηλαδή περιοριζόμαστε μόνο στην φορολογική εποπτεία, που είναι φυσικά ένα πολύ βασικό και αποφασιστική σημασία στοιχείο, αλλά δεν είναι και το μοναδικό. Γιατί νομίζω ότι και η ίδια η Επιτροπή που εισήγε το θέμα της, ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μιλά για απαράβατους όρους οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τα εθνικά σχέδια ή προγράμματα αναθεώρησης με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ένας επικορικός χαρακτήρας των εθνικών προϋπολογισμών. Μέσα στα πλαίσια αυτού του συμπληρωματικού χαρακτήρα και του οριζόντιου χαρακτήρα των φορολογικών, εποπτικών πολιτικών και των άλλων πολιτικών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα μέσα που διαθέτουμε και την εθνική συνιστόσα. Θα πρέπει λοιπόν να εντάξουμε αυτό το μέσο σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Νομίζω όμως ότι δεν αρκεί μέσα στα πλαίσια της εμβέλειας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα έπρεπε να ασχολείται με όλες αυτές τις πολιτικές. Δέχομαι ορισμένες πτυχές της έκθεσης, αλλά θα πρέπει να μιλάμε για έναν ειδικό κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και όχι για ένα ειδικό άρθρο το οποίο εντάσσεται στην έκθεση Wortman Call. Ευχαριστούμε κυρία Γκουαλτιέρη. Ο κύριος Ντάφ έχει το λόγο. Είναι περίπλοκο το ζήτημα και οφείλω να ομολογήσω ότι αδυνατό να κατανοήσω έστω και λίγο τη σχέση ανάμεσα στην έκθεση Μπερές και το πακέτο των έξι οδηγιών. Το εξάμεινο εμφανίζεται ως ιδέα σε διάφορα από τα έξι σχέδια. Δεν πρόκειται μόνο δηλαδή για την έκθεση Βορτμανκόλ που αναφέρεται το εξάμεινο και ο κύριος Γουαλτιέρη έχει δίκιο βεβαίως πως δεν πρόκειται μόνο για τον έλεγχο της ε, ε, δημοσιονομικής ε, πειθαρχίας. Πρόκειται για την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας Αφήστε που δεν σε, ε, δεν νομίζω ότι ό,τι γράψει η κυρία Μπερές μέσα στην έκθεση της ε, σχετικά με αυτό το θέμα ε, θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας. Πιστεύω πάντως πως θα έπρεπε να αναρωτηθεί η Επιτροπή μας για τη σχέση αυτής της έκθεσης με το πακέτο των έξι αν υπάρχει κάποια τέτοια. Ο, ο κύριος Χέφνα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι λίγο το ίδιο με το μηχανισμό σταθερότητας. Προσπαθούμε να ε, πετύχουμε πάρα πολλά με όσο γίνεται λιγότερα μέσα και λιγότερο μοχλό. Και εγώ έχω την εξής ανησυχία. Το μοχλό αυτό δεν το χρησιμοποιούμε σωστά ούτε σε εκείνη τη θέση ε, που θα είναι αρκετά σταθερός και αρκετά βαθιά για να μπορούμε να κινήσουμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, είτε όλα αυτά που γίνονται με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και συνδέονται με αυτό δεν τα εννοούμε σοβαρά, είτε αν τα εννοούμε σοβαρά και θέλουμε να είναι ένα ουσιαστικό ε, στοιχείο συντονισμού των οικονομικών μας πολιτικών, δηλαδή και οικονομικά και δημοσιονομικά ε, στο μέλλον να λειτουργεί, χρειάζεται μια πιο γερή νομική βάση και μια πιο στιβαρή για να μπορεί να σηκώνει περισσότερο βάρος. Συμφωνώ πολύ με τον Γκολτιέρη. Χρειάζεται ξεχωριστός κανονισμός που να μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε ακριβώς ε, τα πράγματα και να λέμε τι εννοούμε με τη διακυβέρνηση. Να είναι γερή η επιφάνεια που σηκώνει όλα αυτά τα θέματα και νομικά και πολιτικά δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε. Διότι αν θέλουμε πραγματικά αποτελεσματικό συντονισμό και τον πετύχουμε, αυτό θα έχει επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, στις πολιτικές στο ιστορικό των κρατών μελών και θα τεθεί το θέμα της νομικής βάσης. Δεν θα είναι ασήμαντο με ποια νομική βάση γίνονται όλα αυτά, διότι θα προκληθούν διαμαρτυρίες κλπ. Έχω λοιπόν μια ανησυχία, γιατί έχω την εντύπωση ότι, πώς να το πω, και πάλι προσπαθούμε να συνενώσουμε ε, με έναν τρόπο τεχνικό. Ε, χτίζουμε ε, πάνω στην άμμο, αλλά θέλει πολύ γερά θεμέλια για να σταθεί αυτό το σπίτι και δυστυχώς δεν το βλέπω. Θα ήθελα ο εισηγητής να λάβει το λόγο, να μας πει τι σκέφτεται. Η πλέον δύσκολη πτυχή της έκθεσης αυτής και της έκθεσης της κυρίας Μπερές είναι αυτό που υπέδειξε ο κύριος Ντάφη σχέση με το πακέτο των έξι οδηγιών. Όταν προετοίμαζε αυτό το σχέδιο, ακόμη νωρίτερα, έτσι, πριν δηλαδή ε, δούμε ξεκάθαρα ποια ε, θα είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων, υπολογίζαμε στην επιτυχία ε, αυτών για το πακέτο των 6. Είχαμε φανταστεί ότι θα ήταν πιο δύσκολο. Αν υπάρξει συμφωνία για το πακέτο των 6 οδηγιών, ε, θα λέγαμε ότι θα είναι η έκθεση για την οικονομική διακυβέρνηση η πιο ισχυρή και δεν θα χρειαζόταν δική μα ε, γνωμοδότηση. Θα ήταν περίτη. Ήταν δύσκολη η απόφαση τώρα, όμω έχουμε περιέλθει σε πάρα πολύ διαφορετική κατάσταση, διότι ακόμη συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις ε, για το πακέτο των έξι και θέλω να είμαστε συνετοί εξ αρχής. Αυτό που επιθυμώ είναι να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό εξάμεινο αφενός που δεν υπονομεύει τη νομική ε, σαφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη συνδυάσουμε με την νομιμότητα και τον εποπτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου, χωρί όμω να υπονομεύσουμε ε, την νομιμότητα των διαπραγματευτών μα ε, στα πλαίσια του πακέτου των 6. για να μην καταδικάσουμε την πιο φιλόδοξη έκβαση, αν θέλετε, των διαπραγματεύσεων για το πακέτο των 6. Και γι' αυτό ε, πήρα αυτή την απόφαση να είμαι μετριοπαθής ε, μάλλον στη γνωμοδότηση και να περιοριστώ ε, στους κανονισμούς που απαρτίζουν το πακέτο των 6. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Να κάνουμε την συζήτηση, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις για το πακέτο των 6 και κατόπιν να λάβουμε την απόφαση και σε συνδυασμό με την θέση που θα τηρήσουν οι διαπραγματευτές μας, οι οποίοι διαπραγματεύονται στα πλαίσια της συναπόφαση για το πακέτο των 6 ούτω ώστε να έχουν μεγαλύτερη ισχύ εκείνοι. Να είμαστε λοιπόν διαλλακτικοί, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, με τις διαπραγματεύσεις, να διευκρινίσουμε ότι ακριβώς ε, θέλουμε, αλλά κυρίως να ενισχύσουμε τη θέση των διαπραγματευτών μας ε, για το πακέτο των έξι, χωρίς όμως να διαχωρίζουμε πλήρως αυτά τα δύο ζητήματα, γιατί έτσι υπονομεύουμε την νομιμότητα των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως είμαι ανοιχτό. αν θέλετε ένα διακριτό κανονισμό για να ενισχύσουμε την ιδέα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ε, και να ε, βελτιωθεί ε, η κατάσταση ως προς την νομική ασφάλεια στην ένωμη τάξη της Ένωσης, ναι, να το συζητήσουμε. Αλλά σήμερα, όπως έχει η κατάσταση, νομίζω ότι θα ήταν πιο σόφρο στις αρχές Σεπτεμβρίου να επανέλθουμε και να ενισχύσουμε τη θέση των διαπραγματευτών μας για το πακέτο των 6. Αυτή είναι η δική μου εισήγηση, αλλά είμαι ανοιχτός σε προτάσεις και αν καταλήξουμε στο ότι για να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική ισχύ των συναδέλφων μας πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να ακολουθήσω κι εγώ αυτή τη γραμμή, αλλά ε, να σας πω επίσης ότι πριν από λίγες εβδομάδες ε, ειλικρινά φαινόταν ότι θα ήταν περιττή η γνωμοδότηση. Αν ε, ήταν να ληφθούν οι αποφάσεις δηλαδή, για την οικονομική διακυβέρνηση, εμείς θα βρισκόμασταν σε μια θέση όπου θα υπονομεύαμε τη δική μας την νομιμότητα, γιατί εμείς που είμαστε οι θεματοφύλακες της όλης διαδικασίας, συγγνώμη, αν περατωθούν οι διαπραγματεύσεις και εμείς είμαστε εκεί πέρα δίπλα ε, και κραδένουμε την σημαία μας ε, με τις φιλοδοξίες μας δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα ε, αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να διαλύσουμε, να διασκεδάσουμε οποιαδήποτε ασάφεια και ανησυχία υπάρχει γιατί υπάρχει παρανόηση και αφήστε δεν μιλάω καν για την παρανόηση στα μυαλά των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τέλο πάντων, ο βασικό στόχο μα είναι να ενισχύσουμε τη θέση των διαπραγματευτών και να μεριμνήσουμε ώστε ο επιπτικό ρόλο του Κοινοβουλίου και η δημοκρατική νομιμότητα τη όλη διαδικασία να κατοχυρωθούν ε, οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Χέφνερ έχει ζητήσει. Ναι, ναι, μία σύντομη ερώτηση έχω και να κάνω και μία σύντομη παρατήρηση σε σχέση με αυτά που ακούσαμε. Πότε αναμένεται η γνωμοδότηση, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για μας, μέχρι πότε πρέπει να αποφασίσουμε, μπορείτε να μου το πείτε. Ήδη είχαμε δεικτικές ημερομηνίε, αλλά καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να τις δούμε με αρκετή ευελιξία. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη Τσαρκόφσκη. Μιλήσαμε για 31 Αυγούστου μέχρι τις 12 το μεσημέρι για υποβολή τροπολογιών και να ψηφίσουμε στις 19 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Τσαρσκόφσκι θα μας πει αν είναι δυνατόν να ψηφίσουν. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Ήθελα να κάνω και μία παρατήρηση. Συμφωνώ ε, απολύτως μαζί σας να μην παρέμβουμε τώρα στις δυσχερέστατες αυτές τις διαπραγματεύσεις με τρόπο που να τις υπονομεύσουμε, να τις βλάψουμε. Ε, όμως ταυτόχρονα έχουμε και ένα ρόλο να διαδραματίσουμε, έχουμε ένα καθήκον, μια αποστολή. Ε, το Κοινοβούλιο και ειδικότερα η Επιτροπή μας ε, είναι αυτή που θα πει ότι ή δυνατόν χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη νομική βάση, αλλά εγώ δεν θα ήθελα απλώ να παρακολουθώ τις διαπραγματεύσεις και να δώσω τη συγκατάθεσή μου. μα ζητείτε η γνώμη μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε λίγο μεγαλύτερη πυγμή. Όχι με τρόπο ώστε να βλάψουμε ε, τελικά τις διαπραγματεύσεις, ε, μόνο να εκφράσουμε σαφέστερα την άποψή μας. Και καταλαβαίνω αυτά που είπατε και ο Ρομπέρτο Γκουαλτιαρή και εσείς ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση κινείστε. Ο κύριο Γκουαλτιέρη θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι κατανοώ την επιχειρηματολογία τακτική υφή του κυρίου Τσαρκόφσκι. Αλλά κάτι έχει αλλάξει, όπως είπε και ο ίδιος. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από μία φάση όπου θεωρούσαμε ότι το τρένο δεν έχει φτάσει στον προορισμό του και πέρα από θέματα ουσίας ως προς την ε, ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το Συμβούλιο μπορεί να δεχτεί ορισμένα θέματα που έλαβαν υπόψη οι εισηγητής. Έτσι ανοίγει το παιχνίδι. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άμεσο αίσιο πέρας. Γι' αυτό ο ρόλος της ΑΦΚΟ ε, γίνεται πιο δεσμευτικός. Δηλαδή να επαναφέρουμε το τρένο στη σιδηροτροχιά του. Γιατί το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα έπρεπε να έπεται του, του πακέτου έξι οδηγιών. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ε, θα, τι κατεύθυνση θα πάρουν οι διαπραγματεύσεις. Και ίσως θα έπρεπε να ασκήσουμε το ρόλο μας γνωρίζοντας ότι αυτά που λέμε εμείς δεν είναι και θέσφατα. Έχουμε όμως από, πλευράς, ε, από θεσμικής πλευράς να γνωμοδοτήσουμε. και μετά μπορεί να αποφανθεί κανείς διαφορετικά. Αλλά θα πρέπει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να κάνει ορισμένες υποδείξεις έτσι ώστε να ξαναδούμε ε, θέματα που μας διχάζουν. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτό το θεσμικό πλαίσιο και μετά θα δούμε πώς διαμορφώνεται ο ρόλος μας. Αυτό θα γίνει με την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γιατί βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση γιατί δεν γνωμοδοτούμε ως προς το πακέτο έξι οδηγιών, όπου θα ήταν και πιο εύκολο να λάβουμε θέση για να ενισχύσουμε τη θέση μας και να εκφράσουμε και την απόψή μας ως προς το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ε, πρόκειται για δύο διαφορετικές πορείες. Πρώτον, διαπραγμάτευση για το πακέτο έξι οδηγιών και την γνωμοδότηση επί της έκθεσης της Περβάων Περές, που φαινόταν ότι θα έπετε των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε ως προς την έκθεση Μπερές, γιατί δεν θα γνωμοδοτήσουμε ως προς το πακέτο 6 οδηγιών, αλλά ως προς την έκθεση Μπερές. Και μέσω των διαπραγματεύσεων ορισμένα ε, στοιχεία παροπλίστηκαν, δηλαδή δεν ε, μιλάμε για μία πρόταση απόφασης για διοικητικά θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συγχρονίσουμε τις δραστηριότητες. Δεν θα πρέπει να είμαστε ουραγοί και παθητικοί. Θα πρέπει να συγχρονίσουμε τη συλλογιστική μας με αυτά που συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις και με θέματα καθαρά χρονισμού, γιατί θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε στην έκθεση υπερβαονσμπερές. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερη γνώση του θέματος της διαπραγματεύσεις και κατά τα τέλη Αυγούστου να έχουμε μια σαφή θέση που θα συγχρονιστεί με το πακέτο των έξι οδηγιών, αυτή τη διαπραγμάτευση. Ε, είχαμε και ορισμένες προτάσεις της ε, Πολωνικής Προεδρίας, προτάσεις ε, που εκφράστηκαν στην αρχή της Προεδρίας από Τώρα θα έχουμε ένα νέο πακέτο προτάσεων, ακόμα και σε αυτό το διάλειμμα του καλοκαιριού. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε μια θέση αρχής και αν ε, συγχρονιστούμε και με την έκθεση Μπερές και με τη θέση άλλων για να έχουμε έναν ξεχωριστό κανονισμό, εγώ τάσουμε υπέρ. Θα πρέπει να αντιδράσουμε στις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας, να συγχρονιστούμε με την τακτική των διαπραγματευτών και να ενισχύσουμε τη θέση μας. Δεν γνωμοδοτούμε για το πακέτο έξι οδηγιών, αλλά γνωμοδοτούμε για την έκθεση της Περβάνς Μπερές και τις συστάσεις που ενυπάρχουν. Αλλά πολλές έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα, διότι έχει, έχει περάσει, μας έχει προσπεράσει το τρένο του πακέτου των έξι οδηγιών. Νομίζω τα περισσότερα στοιχεία ενυπάρχουν υπάρχουν στην έκθεση. Θα πρέπει να συγχρονίσουμε καλύτερα τα πράγματα μέσω τροπολογιών συμβασμού κατά τα τέλη Αυγούστου. Βεβαίως είναι δύσκολο γιατί έχουμε τις διακοπές που μεσολαβούν. Τουλάχιστον όμως να το ε, αναστείλουμε για τις αρχές Σεπτεμβρίου έτσι ώστε να λάβουμε μία απόφαση για τις αρχές του Σεπτεμβρίου για να ενισχύσουμε και τους διαπραγματευτές για το πακέτο 6 οδηγιών και για την έκθεση Μπερές που θα ψηφιστεί στις 17 Σεπτεμβρίου. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να κρατήσουμε τη, τα τέλη Αυγούστου, 19 Σεπτεμβρίου στη συνέχεια και θα βρούμε μια λύση μέχρι τότε. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι στις 7 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσουμε ε, και θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμού σε μια έκτακτη συνεδρίαση στις 7 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια στις 19 ε, Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσουμε από τις 3 μέχρι τις 6.30 και στη συνέχεια θα συνεδριάσουμε στις 5 Οκτωβρίου 2011 από τις 9 έως τις 12.30. Έληξαν οι εργασίες μας. Σας εύχομαι καλές διακοπές. Ο κύριος Νταφ. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή Υπάρχει μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Μάλλον, από όσο γνωρίζω, όλες είναι έκτακτες. Στις 7 Σεπτεμβρίου. Στις 7 Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι. Από πότε μέχρι πότε είπατε, 7 Σεπτεμβρίου. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Από τις 12.30 μέχρι τις, 15 ε, και, μέχρι τις 1 ε, και 15, με συγχωρείτε. Δηλαδή 3 τέταρτα από τις 12.30 στις, στις Βρυξέλλες, 12.30 με 1 και τέταρτο στις 7 Σεπτεμβρίου. Νταφ. Από τις 12.30 μέχρι τη μία και τέταρτο, στις 7. Ναι, ακριβώς, τρία τέταρτα, για τρία τέταρτα, στις 7 Σεπτεμβρίου. Εντάξει. Ξαναρχίζουμε με τους συντονιστές, επαναλαμβάνουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών